Κυρίε και κύριοι, κηρύσω την έναρξη, την έναρξη της συνεδριάσεως μας που διακόπτει χθες. Καλημέρα σας. Και περνάμε στο πρώτο σημείο της τη διάταξης που είναι η δήλωση του Συμβουλίου καθώς και της Κομισιόν για τα μέτρα που έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων του ρεύματος μετανάστευσης που προέκυψε από τον πόλεμο της Συρίας. Δίνω καταρχήν το λόγο στον εκπρόσωπο του Συμβουλίου, τον κύριο Λεσκοβίτσιους. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Καλημέρα σας κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη. Κατά τα τελευταία χρόνια έχουμε δει πολλά σημαντικά γεγονότα στην Συρία, τραγικά γεγονότα, αλλά τώρα η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη. Ο αριθμός των προσφύγων